θα φέρουν πραγματικές αλλαγές και θα κλείσουν το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα η σε διάταξη προβλέπει την ε, συζήτηση της εκθέσεως του κύριου Τριανταφυλλίδη, ενίσχυση της αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στον τομέα του ασύλου. Κύριε Τριανταφυλλίδη, Έχετε το λόγο. Είστε εδώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου μας απασχολούν εδώ και χρόνια και όπως όλα δείχνουν η φετινή χρονιά θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του και συνεπώς την έναξη μια νέα περίοδου. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου δεν θα είναι αντάξιο των αρχικών μα προσδοκιών παρά τα αυτά ελπίζουμε πως θα γίνουν έστω κάποια θετικά βήματα και ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα έστω και σταδιακά. η παρούσα έκθεση εντάσσεται σε αυτήν ακριβώς τη σταδιακή λογική. ως κοινοβούλιο στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα προς την ευρωπαϊκή επιτροπή και τα κράτη μέλη όσον αφορά τις προσδοκίες μας σχετικά με την ενίσχυση της αλληλεγγύης στον τομέα του ασύλου εντός της ευρωπαϊκής ένωσης. μέσω αυτού του κειμένου έχουμε καταφέρει να μεταφράσουμε σε συγκεκριμένους όρους την αφηρημένη έννοια της αλληλεγγύης τονίζοντας τη σημασία της δίκαιης κατανομής των ευθυνών μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Τώρα περιμένουμε από την Επιτροπή να μας διαβιβάσει σχετικές νομοθετικές προτάσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο που δεσμευτήκαμε να αναλάβουμε ήδη από το 1999. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου για την εξαιρετική συνεργασία στο φάκελο αυτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Merci Monsieur Trentafilides. Ε, nous passons à la procédure 4. Περνάμε στη διαδικασία 4 Ο κύριος Παπανικολάου, πρώτος ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ε, εκ μέρους της ομάδας μας, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της κοιόδους εισηγήτριας της κυρίας Χολμάιερ και εμού προσωπικά θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή μας για την πολύ καλή έκθεση, να τονίσω ότι ήταν πολύ σημαντική η συζήτηση που διεξήχθη κατά τη διάρκεια ε, της ε, προεργασίας και της σύνταξης εκθέσεως αυτής, τη στιγμή που προχωρά η διαπραγμάτευση για το πακέτο ασύλου που όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να το ολοκληρώσουμε ε, μέσα σε ε, δύσκολα χρονικά περιθώρια μέχρι το τέλος της χρονιάς αυτής. Η έκθεση αυτή μας έδωσε ευκαιρία να αναπτύξουμε πιο ανοιχτά τις σκέψεις μας, να καταθέσουμε προτάσεις και ιδέες και πραγματικά νομίζω ότι η έκθεση αυτή και μετά την ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης θα αποτελεί σημείο αναφοράς ό,τι αφορά, ε, όπως σωστά ανέφερε και ο εισηγητής, τα προβλήματα που έχει ε, το κοινό πακέτο ασύλου την ανάγκη για περισσότερη αλληλεγγύη την ισότιμη κατανομή των βαρών. χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου χρειαζόμαστε υψηλά επίπεδα προστασίας όλα αυτά αναφέρονται στην έκθεση και θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον εισηγητή και βεβαίω όλες τις πολιτικέ ομάδε για την προσπάθεια που έγινε. Ε, Σα ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Ρωμέβα. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή. Μεταξύ άλλων, η έκθεση διασφαλίζει τον, την καλή λειτουργία του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό όπω η σημερινή συγκυρία. Το ακούσαμε και πιο πριν. Ο αριθμός των ατόμων που αποβιώνουν όταν προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη με το ταξίδι που κάνουν. Βλέπουμε πάρα πολύ καλά όπως, η έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων οδηγεί στην άρθρωση λόγου όπω τη χρυσή αυγή στην Ελλάδα που ανησυχεί ιδιαίτερα ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό το γεγονό. Το θέμα τη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών είναι υποχρέωση, όχι μόνο ανθρωπιστική, αλλά και ανθρωπιστική ευθύνη και υπευθυνότητα, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε σχέση με τι χώρε μα που πρέπει να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνε του. Είναι πάρα πολύ αναγκαία τα μέτρα που προτείνονται από την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Η κυρία Μαζασκούκοβιτς, παρακαλώ. 670. Mm-hmm. Όχι, δεν είναι εδώ η κυρία Μπασέσκου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Το πρόβλημα του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα πολύ ευαίσθητο Υπάρχουν ακόμα πάρα πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα αιτήματα από τους ετούντες άσυλο. Μπορούν να επιληθούν μόνο με μεγαλύτερη έκφραση αλληλεγγύης από τα κράτη-μέλη. Η δημιουργία της υπηρεσίας για το άσυλο έχει ακριβώς αυτό το στόχο. Να μπορέσει να αρθρώνεται σωστά αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Η Ρουμανία αντελήφθη την ανάγκη να συνεργάζεται με εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό ετούντων άσυλο. Η Ρουμανία όμως δεν έχει τόσο τέτοιο μεγάλο αριθμό. Η χώρα μου παρόλα αυτά έχει αντιληφθεί την ανάγκη να συνεργάζεται με τις άλλες χώρες για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Στις μελλοντικές προοπτικές το Ταμείο για το Άσυλο και την Μετανάστευση θα οδηγήσει στην στο καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Φρασίκοβα. Ευχαριστώ κυρία Φρασίκοβα, Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να ολοκληρώσει μέσα στο 2012 το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου με την κοινωτική προστασία, ενιαίες διατάξεις και ισότιμη παροχή διεθνούς προστασίας. Είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει το σύστημα αυτό. Οι μεταναστευτικές ροές συχνά είναι μικτές, περιλαμβάνουν δηλαδή και μετανάστες και τούντες άσυλο αλλά και ανηλίκους ασυνόδευτους. Αυτές οι μεταναστευτικές ροές με τις ιδιαιτερότητές τους πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά περίπτωση. Τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να χειριστούν και να επεξεργαστούν όλες τις αιτήσει ασύλου και πρέπει να βρούμε καλύτερες λύσεις, να, δώσουμε, να εξασφαλίσουμε καλύτερη κατανομή αρμεδιοτήτων και απαιτείται βέβαια η ενίσχυση της τεχνικής συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τσόρον παρακαλώ. είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μάλτα η ελλάδα η ιταλία στη λαμπεντούζα κτλ. αλλά δεν είναι τόσο γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αλλά από κοινού το πρόβλημα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ένα θέμα λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή πολιτική. Σημειώνω εδώ με ικανοποίηση το ότι πολλοί χρησιμοποιούν τον όρο Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και χρειάζεται καλύτερος έλεγχος, ίσως και κοινή υπηρεσία φύλαξης των συνόρων, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που δημιουργείται με τους πρόσφυγες και τους παράνομους μετανάστες, αλλά σεβόμενοι φυσικά την αξιοπρέπειά τους. Ευχαριστώ κύριε Σπάσκο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επιτροπέ, όλο και περισσότεροι είναι οι μετανάστες που προξένησε η Αραβική Άνοιξη και βλέπουμε ότι αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία η πολιτική του ασύλου. Τα νοτιότερα κράτη της Ευρώπης είναι εκείνα τα οποία πλήττονται περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα στη συνεργασία και με τα άλλα κράτη-μέλη. Απλή λύση ε, που ενδεχομένως χορηγείται δεν δίνει πάντοτε τα απαιτούμενα αποτελέσματα και την επιτυχία που απαιτείται. Οι μετανάστε αυτοί έρχονται συχνά στην Ευρώπη γιατί απλώς αναζητούν καλύτερε συνθήκε ζωή. Γνωρίζουν ότι οι πρώην απεικιοκρατικέ δυνάμεις των οποίων γνωρίζουν και τη γλώσσα μπορούν να του επιτρέψουν ε, λόγω τη γλώσσα, να ενσωματωθούν πιο εύκολα στην ε, κοινωνία. Έτσι λοιπόν ένα Αλγερινό ή ένα Ινδός ο οποίο έρχεται στη Γαλλία ή τον Εμένο Βασίλειο μπορεί να θεωρεί ότι θα ενσωματωθεί καλύτερα αλλά αν πάει στη Ρουμανία ή σε κάποια άλλη χώρα χώρα ε, τη οποία γνωρίζει τη γλώσσα αντιμετωπίζει μεγάλε δυσκολίε. Και εκεί δεν επιλύονται εύκολα τα προβλήματα. Για να αντιμετωπιστούν λοιπόν καλύτερα αυτέ οι καταστάσει, θα πρέπει να χορηγείται η δυνατότητα στον ετούντα το άσυλο ε, τη επιλογή σε ποια χώρα θέλει να ζήσει ώστε να μπορεί να σωματωθεί καλύτερα στην κοινωνία. Ευχαριστώ κύριο Νικολάση για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, το κοινό σύστημα ασύλου πρέπει να ολοκληρωθεί το μέσα στο 2012 μέσα από μια νέα ε, επεξεργασμένη μορφή. Πρέπει το σύστημα αυτό να εξασφαλίζει για όλα τα κράτη-μέλη ένα κοινό προνομαστή, μια κοινή βάση εργασίας και βλέπω ότι υπάρχουν χώρες που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα ροές μεταναστευτικές από τη Βόρεια Αφρική κυρίως, η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ιταλία, αλλά και άλλες χώρες όπως η δική μου πατρίδα αντιμετωπίζουν νέες ροές μεταναστών που πλέον δεν αντιμετωπίζουν τη χώρα μας σαν ε, χώρα μόνο διέλευσης αλλά και σαν χώρα προορισμού. Υπάρχουν πολλοί μετανάστες δηλαδή που ε, θέλουν να εγκατασταθούν στη Σλοβακία. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος ε, πρέπει να σας πω ότι έχει, ε, για το ότι έχει η πατρίδα μου εισαγάγει ένα σύστημα ανθρωπιστικό για το άσυλο, ένα φιλόξενο σύστημα, προσφέρει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και καλές δυνατότητες για ενσωμάτωση στην κοινωνία και ήθελα να υπογραμμίσω αυτή τη διάσταση. Ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στον κύριο Επίτροπο. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, να ευχαριστήσω τον κύριο εισηγητή, τον κύριο Τριανταφυλλίδη και όλα τα μέλη τα οποία πήραν μέρος στην προετοιμασία της έκθεσης. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανάπτυξη της ε, εσωτερικής αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του ασύλου. Η αρχή της αλληλεγγύης φυσικά συμβαδίζει με την αρχή της ευθύνης όσων εμπλέκονται. Ο χώρος στα πλαίσια του οποίου θα αναπτυχθεί η αρχή της αλληλεγγύης έχει επιβεβαιωθεί και η ε, κάθετη και η τεχνική συνεργασία θα πρέπει να συμβαδίζουν με την νομοθετική εναρμόνιση. Η οικονομική αλληλεγγύη μέσω στενότερης εταιρικής σχέσης είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει όπως επίσης και η σωστή διανομή των πιστώσεων στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτούς που αιτούνται ασύλου. Η δράση μας στον τομέα της ελληνικής θα πρέπει να είναι πλήρης και ισορροπημένη, η αμοιβαία στηρίξη θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο του χώρου αυτού και στον τομέα της επανεγκατάστασης και στον τομέα της εύρυθμης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συνολικά Συστήματος. Η αλληλεγγύη και το άσυλο δεν αφορούν κάτι το κατεπήγον ή μία θα έλεγα αντίδραση σε ένα απλό φαινόμενο. Η αλληλεγγύη πρέπει να χαρακτηρίσει την καθημερινή πρακτική στα κράτη-μέλη υποστηρίζοντας σαν παράδειγμα τις προσπάθειες επανεγκατάστασης όχι μόνο γιατί το θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται πολύ στην επικαιρότητα αλλά γιατί επειδή έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Τον προηγούμενο Μάρτιο στην ετήσια έκθεση εμείς για τη μετανάστευση και, και το άσυλο ή μάλλον τον επόμενο Μάρτιο θα δημοσιεύσουμε τα επόμενα στοιχεία τα οποία θα έχουμε συγκεντρώσει περιγράφοντας την κατάσταση. Ασκείται κριτική στην έκθεση σε σχέση με τον αφορμαγή του κανόνα του, της ρυθμίσεως του Δουβλίνου και ε, προτείνεται ένα νέο σύστημα για την ανακατανομή των ετούντων άσυλων το σύστημα του Δουβλίνου δεν είναι ιδανικό πράγματι λόγω της γεωγραφικής του θέσης ορισμένες χώρες υφίστανται πάρα πολλές δυσανάλογες πιέσεις. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Τα κράτη-μέλη χωρίς εξωτερικά σύνορα επηρεάζουν όμως και αυτά μερικές φορές από δυσανάλογες μεταναστευτικές ροές. Βέβαια τα επίπεδα αντιμετώπισης του προβλήματος είναι άνισα σε διάφορες χώρες μεταξύ τους. Αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της μεταρρύθμισης ε, της, ε, ε, του κανονισμού του Δουβλίνου και του CACS. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Ντάλι, λέει η Πρόεδρος. Περνάμε στο επόμενο σημείο την συζήτηση για την φαρμακοεπαγρύπνηση, κοινή συζήτηση για την έκθεση της κυρίας Λίντα Μακάβαν. Η μία έκθεση αφορά την τροποποίηση της οδηγίας και η άλλη την τροποποίηση του κανονισμού. Ξεκινώντας θα δώσω το λόγο στην κυρία Μακάβαν για τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.